So thank you. Those leaving the room, please. Σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ αποχωρήστε ησύχως και σιωπηρά. That we can proceed to the second panel. With no recess. We thank you. Μπορούμε λοιπόν, αν ευδιακοπής, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ευρωπαϊκή Ένωση επαν... Πολιτική Επανεισδοχή και οι συνέπειες για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To introduce the panel. We're going to be talking here. Λοιπόν, παρουσιάζω το πάνελ. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το πάνελ στην συνεδρίαση την κοινή της Επιτροπής των ε, εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Η πολιτική αυτή επανιστοχή είναι ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να ενισχύσουμε την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και θέλουμε να τονίσουμε ότι η ανάπτυξη αυτή τη πολιτική σε επίπεδο ευρωπαϊκού επίπεδου θα επιτευχθεί μονάχα με μια συνολική προσέγγιση στις πολιτικές μετανάστευσης. για την πολιτική αυτή επανεισδοχή είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι πολύ σημαντικές, για την ευρωπαϊκή πολιτική. Όλα αυτά εμπλέκουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από τότε που τέθησε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ξέρετε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την αρμοδιότητα του να δώσει την σύμφωνη ή ασύμφωνη γνώμη του βάσει του άρθρου 18 σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες αυτού του χαρακτήρα και έχουμε το τελικό λόγο σε οποιαδήποτε συμφωνία που έχει να κάνει με επανεισδοχή μέσα στην πολιτική μετανάστευσης. Το πάλι ποτέ, το 2010, όταν συζητούσαμε την πρώτη συμφωνία επανεισδοχής, υπήρξε μια δήλωση της Κομισιόν που προσθέθηκε ως παράτημα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέγον η Κομισιόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τηρηθεί ενήμερο σε τακτά διαστήματα σε σχέση με τη σύναψη συμφωνιών επαρισδοχής μέσα στο πλαίσιο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορα επίπεδα θα συμμετέχει στη συνεδρία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την άσκηση των εξουσιών σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου για τις συμφωνίες επανιστοχής, η συνεργασία αυτή θα εφαρμόζεται με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξασφαλίσει και τον απαραίτητο έλεγχο και προφανώς θα έχει τη συνέπεια της βελτίωσης της ουσίας της πολιτικής επανεισδοχής ως σύνολο. Και γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά για την επόμενη ώρα. Πώς θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικότερο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε προσθέμενη αξία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την ε, αναθεώρηση της πολιτικής επανιστοχής ως τμήμα της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Δίνω καταρχήν το λόγο στον κύριο Jean-Pierre Κασαρίνο ως Διευθυντή της πλατφόρμας για την ε, ε, επανεισδοχή και την ε, μετανάστευση στο Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Ευχαριστώ κύριε Δαγκυλάρ, θα μιλήσω γαλλικά. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, είναι μεγάλη, μια μεγάλη τιμή που λαμβάνω εδώ το λόγο ενώπιόν σας και ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους. Η σύντομη παρέμβασή μου αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επανεισδοχών και την εφαρμογή του ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια είναι σωστό που μιλάμε για σύστημα διότι υπάρχουν πάρα πολλές συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τα κράτη-μέλη της Ένωσης και την Ένωση την ίδια κάθε αυτήν. Βέβαια δεν μπορώ σε 10 λεπτά να σας αναφέρω όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του συστήματος που συνεχώς επεκτείνεται από τα κρατικά συμφέροντα μέχρι άλλα συμφέροντα. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο θέμα της, του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπως είπε ο κύριος Δαγκυλάρ, από τότε που τέθηκε ενισχύει η συνθήκη του Αμστελοδάμου η Ένωση έχει δικές της δικαιοδοσίες ως προς τις επανεισδοχές και η συνθήκη της Λισαβόνας αργότερα τις επέκτηνε περαιτέρω. Βέβαια, η ύπαρξη μιας ε, κοινή δικαιοδοσίας κρατών και ένωσης δεν είναι προβληματική αν την διέπει η αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας Το το αναφέρει και η συνθήκη. Την αναφέρει και η συνθήκη. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου και αξιολόγηση για την εφαρμογή και πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης. Δηλαδή το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των προσώπων ε, και των μειονοτήτων και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όπως στο άρθρο 2 και στο άρθρο 6 της Συνθήκης της Ένωσης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι, ως προϋπόθεση ότι υπάρχει κάποια σύγκληση μεταξύ των προτεραιοτήτων των χωρών μελών και εκείνων της Ένωσης. Πράγμα στο οποίο θα επανέλθω αργότερα αλλά πολύ σύντομα. Για ως προς τους μηχανισμούς τώρα της εποπτείας ή του ελέγχου. Θα ήθελα να επιμείνω ότι οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συγκεκριμένη εφαρμογή τους είναι δικαιοδοσία των χωρών μελών στα πλαίσια των πρωτοκόλων, διμερών πρωτοκόλων εφαρμογής που έχουν υπογραφεί μεταξύ το, της κάθε χώρας και τρίτων χωρών που έχουν τέτοια συμφωνία με την Ένωση για τις επανεισδοχές και διέπονται από την Μικτή Επιτροπή Επανεισδοχών. Αυτή η Μικτή Επιτροπή Επανεισδοχών είναι ο χώρος όπου ελέγχεται η εφαρμογή των συμφωνιών αυτών. Αλλά προς στιγμήν το μόνο που κάνει είναι να ασχολείται με τεχνικά θέματα για την εφαρμογή της συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτή η Μικρή επιτροπή επανεισδοχών πρέπει να διαθέτει και μία πρόσθετη δικαιοδοσία όπου οι αρμόδιοι παράγοντες να μπορούν να επαληθεύουν τις αληθινές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που υποβάλλονται στην επανεισδοχή. κάτι που είναι απαραίτητο, πόσο μάλλον που η Ένωση έχει υπογράψει συμφωνίες, συμβάσεις επανεισδοχής με χώρες που δεν έχουν συνυπογράψει και τη συνθήκη της Γενέβης του 1951 για τους πρόσφυγες, όπως το Πακιστάν. Και αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις ως προς το σεβασμό και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις εκδόσεις ανθρώπων που περνούν από το Πακιστάν. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνίες με τρίτε χώρες που έχουν υπογράψει αυτές τη συνθήκη τη Γενέβη, αλλά που δεν έχουν σύστημα χορήγηση ασύλου, όχι αποτελεσματικό τουλάχιστον όπως η Ουκρανία που είναι υπόδειγμα σε αυτή την περίπτωση αρνητικό. Η πάτη αρμοστία του ΟΗΕ το τόνισε αυτό, τον κίνδυνο δηλαδή να υπάρξουν ασυνήθεις διαδικασίες επανεισδοχής ή από την Ουκρανία. Υπάρχουν λοιπόν τρίτες χώρες που το, η Πάτια Αρμοστία δεν τις θεωρεί σίγουρες, όπως την Σερβία. Έχουν υπογραφεί επίσης συμφωνίες με τρίτες χώρες όπου είναι προβληματική η ύπαρξη πολλών απατριδών, όπως το Κοτσιφοπέδιο. όπου έχουν σημειωθεί επανεισδοχές. Υπάρχει εδώ ένα εφέ ντόμινο, αλλά ο νόμος πάντοτε τιμωρεί την παράνομη διέλευση συνόρων. Το πρόβλημα λοιπόν, τα προβλήματα είναι πολλά και η οξύτητά τους απαιτεί να αντιμετωπιστούν με τρόπο πολύ διαφορετικό από την απλή ελαστικότητα που εφαρμόζεται μέχρι τώρα και που είναι η βάση της εφαρμογής των συμφωνιών. Πόσο μάλλον που η χάρτα των θεμελιωδών από τότε που τέθηκε ενισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας ε, συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη και έχει την ίδια αξία και σημασία. Το άρθρο 17 της συνθήκης λοιπόν λέει ότι ένας από τους στόχους της Ένωσης είναι τελείως ανεξάρτητα να έχει επιτροπή την ε, εφαρμογή της συνθήκης. Εδώ αυτό σημαίνει και ένα καθήκον εποπτείας. Άρα απαιτείται η δικαιολόγηση οποιασδήποτε επανεισδοχής εφόσον συμπεριλαμβάνει και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και δικαιολόγηση, εξήγηση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται κάθε φορά για να ταυτιστούν οι τρίτες χώρες με τις οποίες οι συμφωνίες για επανεισδοχή μπορεί να συμφωνηθούν στο μέλλον. Γνωρίζω λοιπόν ότι τα κριτήρια αυτά έχουν ήδη καθοριστεί από το 2002, αλλά η εποχή εκείνη ήταν πολύ συγκεκριμένη φάση στην οικοδόμηση της Ένωσης. Μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας και την συμπερίληψη της χάρτας στο θεμελιώδες δίκαιο της Ένωσης πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά τα κριτήρια. Δεύτερο θέμα η σύγκληση των προτεραιοτήτων που είναι και αυτή η απαραίτητη προϋπόθεση για μια ειλικρινή συνεργασία μεταξύ χωρών μελών και Ένωσης. Όπως ξέρετε σε διμερές επίπεδο τα κράτη πάντοτε συνεργάζονται για τις επανεισδοχές μεταξύ τους. Και αυτή τη διμερή συνεργασία η Κομισιόν την έχει προβλέψει από καιρό. Η διμερής λοιπόν συνεργασία για τις επανεισδοχές ε, προϋποθέτει βέβαια αμοιβέ υποχρεώσεις αλλά πολύ άνισα. Πολλές χώρες έχουν καταφέρει οι διπλωματικές πιέσεις να μην τις πείθουν για σωστή συνεργασία και επίσης οι πιέσεις, τέτοιες πιέσεις να καταλήγουν σε υπονόμευση τη αγώνα καταπολέμησης διεθνούς τρομοκρατίας, παράνομη διέλευση συνόρου, ενεργειακής ασφαλείας κλπ. Έτσι λοιπόν υπονομεύεται η δημιουργία μιας σφαιρικής συνολικής συνεργασίας. Όταν μιλάω για μια πιο διευρυμένη συνεργασία εννοώ ότι οι επανεισδοχές σε διμερές επίπεδο συμπεριλαμβάνονται σε ένα χώρο όπου τα εσωτερικά, τα εξωτερικά, τα εμπορικά συνδυάζονται. Αν λοιπόν η διμερή συνεργασία για τις επανεισδοχές μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σημείο κλειδί, παρόλα αυτά η σχετική της σημασία αξιολογείται πάντοτε από τα κράτη-μέλη με βάση άλλα στρατηγικά κριτήρια που τα θεωρούν πιο για Κίνα. Δεν θα μιλήσω αυτό, άμα θέλετε μετά στη συζήτηση. Πάντως αυτές οι διμερείς ε, συνεργασίες δεν συμφωνούν και πολύ με όσα έχει θεσπίσει η κοινότητα από τη συνθήκη του Αμστελοδάμου και μετά. Διότι όλα υποβάλλονται στο κριτήριο της λεγόμενης αποτελεσματικής συνεργασίας. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο θέμα των επανεισδοχών και στις σχέσεις τρίτων χωρών με την Ένωση. Άλλη πτυχή επίσης που είναι ειδική για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών κυριαρχεί στις ε, σχέσεις με τις τρίτες χώρες ενώ νομίζω ότι η Γενική Διεύθυνση για τις εξωτερικές σχέσεις θα έπρεπε να είναι η αρμοδιότερη για να προωθηθούν, για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι που έθεσε η Ένωση για τις εξωτερικές αυτές σχέσεις. Οι επανεστοχές λοιπόν ακόμη διέπονται από τη λογική της ευελιξίας, της λογικής και δεν συμβαδίζει και πολύ αυτό με τα διεθνή πρότυπα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κινητικότητα είναι κάτι που επικίνδυνο για μερικές χώρες, δηλαδή ενισχύεται έτσι η αυθαιρεσία και θεωρείται η Ευρώπη σαν απλώς ένα απαραίτητο κακό. Άρα η ευελιξία εδώ παίρνουν το προβάδισμα μπροστά στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων για τους αιτητές ασύλου και τους πρόσφυγες και τα δικαιώματά τους. Δεν ξέρω κατά πόσον το διώνυμο εσωτερικές υπηρεσίες και υπηρεσία εξωτερικών δράσεων θα μπορούσαν κάποτε να λύσουν αυτό το πρόβλημα των επανεισδοχών και με ποια πολιτική. Αντίθετα όμως ξέρω ότι οι συμφωνίες επανεισδοχών είτε είναι ευρωπαϊκές είτε είναι διμερείς γίνονται αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής από τις ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνώς και εθνικός και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Στις χώρες της Βόρειας Αφρικής ας πούμε προσέχουν πολύ αυτό το θέμα γιατί από την Αραβική Άνοιξη έχουν σημειωθεί τρομερές παραβιάσεις στην ελευθερία διακίνησης, έκφρασης κλπ. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό εκθέτει κυρίως τους ηγέτες των χωρών αυτών, αλλά ταυτόχρονα και την ίδια την Ένωση στην οποία θέτει καινούργια και ανυπέρβλητα, αν καινούργιες ανυπέρβλητες μέχρι τώρα προκλήσεις. Η πολιτική που εφαρμόζει για τις επανειστοχές δεν μπορεί να συνεχίσει λοιπόν έτσι. Για να καταλήξω λοιπόν θα έλεγα ότι σήμερα υπάρχει, έχουμε ένα κριτήριο που είναι της προστιθέμενης αξίας όπως λένε. Και αυτό από τη συνθήκη του Αμστελοδάμου και μετά. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω χωρίς να με θεωρήσετε πολύ ιδεαλιστή ότι η πιο αξιόπιστη αξία που θα μπορούσε να προβάλλει η Ένωση για τις σχέσεις της με τρίτες χώρες, για τις επανειστοχές, είναι ακριβώς ο έλεγχος του κατά πόσον γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί είναι φανερό ότι ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι ζωτικό, όπως και ο μελλοντικό ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Να, αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μαρίνα Σραμ από τον Διεθνή, Φορε... Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα και εξ ονόματος του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση Θέλω να σας ευχαριστήσω που με έχετε καλέσει να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Ο οργανισμός μας δεν εμπλέκεται στην ε, καταναγκαστική επιστροφή των μεταναστών. Υποστηρίζουμε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν ε, συνάψει συμφωνίες επανεισδοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζουμε επίσης τα θέματα παρακολούθησης της κατάστασης συγκεκριμένων ατόμων μετά από την επανεισδοχή τους. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να σας παρουσιάσω μερικά γενικά σχόλια σε σχέση με τα θέματα αυτά. Όπως είπε ο κύριος Κασαρίνο, η επανεισδοχή είναι ένα διαδικαστικό έργο για να εξασφαλίσει την εφαρμογή μιας απόφασης απέλασης, ώστε ούτω δεν πρέπει λοιπόν αυτό το μέτρο να έχει επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα. και γενικά. Θα πρέπει η συμφωνία αυτή η πανιστοχής να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της χώρας στην οποία επιστρέφεται ο μετανάστης και σε περίπτωση ανησυχιών και ε, ενδιασμών δεν θα πρέπει να, λαμβάνεται, να γίνεται αυτή η διαδικασία επανιστοχής. Αλλά από την άλλη μεριά αυτή η διαδικασία μπορεί να διευκολύνει τις διαδικασίες και φυσικά δεν θέλουμε η απλοποίηση των διαδικασιών να υπερκεράσει την ανάγκη, την να δώσουμε στους ε, ε, κρατούμενους το δικαίωμα να, να έχουν πλήρη πρόσβαση στα δικαιώματά τους πριν από την διαδικασία επανεισδοχής. Πολλές χώρες υποδοχής μπορεί να θεωρήσουν ότι τα άτομα αυτά του ατόμου που υπόκειται σε επανεισδοχή έχουν πράγματι εκτιμηθεί πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως δεν έχουν άλλη πρόσβαση σε διαδικαστικά σε δικονομικά μάλλον δικαιώματα μετά την επανεισδοχή τους. Και τώρα θα ήθελα να περάσω στο θέμα της εποπτείας. Υπάρχουν δύο τομείς εποπτείας για τη διαδικασία επανεισδοχής. Από τη πλευρά πόσο αποδοτικές και πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαδικασίες, αλλά αυτό καλύπτεται κυρίως από τις κοινέ επιτροπές επανεισδοχής. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη μεταχείριση των ατόμων που υφίστανται, που την χάνουν επανεισδοχή. Τι γίνεται πριν και μετά από την επανεισδοχή ο Οργανισμός για τη Μετανάστευση παρακολουθεί περισσότερο το τι γίνεται μετά από, τη μετανα... από την επανεισδοχή. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Καταρχήν τι γίνεται αμέσως μετά την επανεισδοχή. Πώς τα άτομα αυτά τα οποία επιστρέφουν σε μια χώρα ε, αντιμετωπίζονται όταν είναι σε διέλευση, όταν φτάνουν στη χώρα αυτή, αλλά τελικά πόσο βιώσιμη και είναι η επιστροφή τους, τι ευκαιρίες έχουν να επανενσωματωθούν στην κοινωνία όπου έχουν επιστραφεί. Υπάρχουν δύο κατηγορίες τέτοιων ατόμων που θέλουμε να εξετάσουμε λίγο καλύτερα σε σχέση με τις ανάγκες τους. Καταρχήν, οι υπήκοοι της ίδιας της χώρας, αυτό αφορά περισσότερο χώρες όπως είναι η Γεωργία, το Πακιστάν, η Σρι λάνκα Θέλουμε να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι όταν γυρίσουν στη χώρα τους έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία πρέπει να έχουν, στα δικαιώματά τους, μπορούν να έχουν ε, έγγραφα σε σχέση με τις ιδιοκτησίες που έχουν, να ξαναπάρουν τα έγγραφα που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή τους κατάσταση και τα οποία ενδεχομένως τα έχουν χάσει. Πρέπει όμως να δούμε και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι η επανεισδοχή τους με την έννοια ότι αυτά τα άτομα μπορούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους μετά από την επανεισδοχή και επίσης είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τις τοπικές αρχές και να εξασφαλίσουμε ότι έχουν επίγνωση των προβλημάτων τα οποία τίθενται για τα άτομα αυτά και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τα άτομα αυτά μετά την επανεισδοχή τους. Η δεύτερη κατηγορία είναι πολίτες τρίτων χωρών. Είναι ακόμα πιο σημαντικό να εξετάσουμε την κατάστασή τους όταν πρόκειται για χώρες διαδιέλευση όπως είναι η Ουκρανία που αναφέρθηκε προηγουμένως. Εκεί μία από τις μεριμνές μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι έχουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, αλλά αυτό θα καλυφθεί από άλλους ομιλητές. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως παραδείγματο χάρη όταν μιλάμε για επανεισδοχή. Το κύριο ζήτημα είναι να δούμε αν υπάρχει μία πρόσβαση σε μία κατάσταση μόνιμου χαρακτήρα. Θα πρέπει να γίνεται μία επανεισδοχή σε τρίτη χώρα, εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή του στην δικιά τους χώρα. <clears throat> θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην τρίτη χώρα, την τρίτη τη χώρα διέλευσης, αν τα άτομα αυτά έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στην τομική κοινωνία, αν μπορούν να επωφελθούν από διαδικασίες που θα τους δώσουν προσωρινή άδεια διαμονής και πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις άλλες ανάγκες που μπορούν να έχουν. Και τι γίνεται μόλις γυρίσει κάποιος σε στη χώρα επανεισδοχής άμα είναι πολίτης τρίτη χώρα. Θα έχουν δικαίωμα στη διερμηνία, θα του εξηγήσουν τι γίνεται και ποιε είναι οι διαδικασίε σε κάποιε χώρε. Τι θα είναι κατευθείαν σε κράτηση αυτοί οι οποίοι έχουν τύχη επανεισδοχής. επειδή θεωρείται ότι ήταν παράνομοι μετανάστες και πρέπει να τεθούν σε ευαγή σοφρονιστικά ιδρύματα ή χώρους κράτησης. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ανησυχίες σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να τύχουν παρακολούθησης. Αυτό που έχουμε κάνει πρόσφατα είναι ότι μαζί με την Κομισιόν έχουμε εργαστεί σε πιλωτικά προγράμματα τα οποία να ξεκινήσουν είτε στο τέλος του χρόνου είτε στην αρχή του επόμενου έτους και που θα εστιάζουν στην Ουκρανία και το Πακιστάν, δύο χώρες που παραμένουν στο επίκεντρο της παρακολούθησης λόγω ορισμένων προβλημάτων. Και εδώ βρισκόμαστε σε εταιρική σχέση και συνεργασία με την υπάτη αρμοστία για τους πρόσφυγες και με την κοινωνία των πολιτών για να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται μετά την επανεισδοχή. Και να δούμε όχι μονάχα τους ε, υπηκόους αυτών των χωρών αλλά και τους πολίτες τρίτων χωρών που <clears throat> γυρίζουν σε αυτές τις χώρες να παρακολουθήσουμε σε βάθος χρόνου τριών ετών τι γίνεται μετά την επαρισδοχή τους. Και έτσι μπορούμε να έχουμε και κάποια ανάδραση σε σχέση με την ε, μορφή της διακυβέρνησης και να έχουμε τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε κυρία Σραμ. Και τρίτη στη σειρά, κυρία Έλεν Σούπιος Ντέιβιτ, η οποία είναι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες υπεύθυνη για ζητήματα συνόδευτων ανηλίκων και επανεισδοχής. Όπως ε, αναφέρθηκε εκπρόσωπο το ΕΚΡΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο για τους Πρόσφυγες που είναι ένα, μια ομοσπονδία πάνω από 70 μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη που ασχολούνται με θέματα ασύλου. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να αναφέρω την θέση του ΕΚΡΑ σε σχέση με την ε, απέλαση. Προφανώς τα κράτη-μέλη έχουν το κυριαρχικό δικαίωμα να ε, επιλέγουν ποιος ε, εισέρχεται στην επικράτειά τους και άρα το δικαίωμα να ε, απελάβουν. Αυτή στιγμή έχει τηρηθεί η διαδικασία ασύλου, δηλαδή έχει δοθεί η δυνατότητα στο πρόσωπο να εκφράσει το αίτημα ασύλου του και αυτό έχει εξεταχθεί εξατομικευμένα και δεόντως. Η επανεισδοχή είναι ένα εργαλείο το οποίο η συμφωνία επανεισδοχής είναι ε, απλώς ε, ένα εργαλείο που διευκολύνει τις απελάσεις και ως εκ τούτου δεν είναι από μόνο του μια ε, συμφωνία που παραβιάζει να ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής θέτει ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολύ συχνά αυτά τα θέματα δεν την χάνουν συζήτησης Γι' αυτό πρέπει να πω ότι είμαι και ευτυχής για τη σημερινή συζήτηση. Ποιο είναι το πρόβλημα από την, κατά την άποψη του ΕΚΡΕ. Η ουδετερότητα και η σύναψη αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής βασίζεται στην παραδοχή ότι η ε, διαδικασία θα είναι δίκαιη και δεν θα σημειωθούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της επανεισδοχής. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει να κινδυνεύσει ακόμα και η ζωή ανθρώπων. Ε, συμπληρωματικά προς εκείνα που είπε ο κύριος Κασαρίνο, που ήδη ανέφερε πολλά θέματα και προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμείς θα θέλαμε κυρίως να αναφερθούμε στην ε, ανεπάρκεια της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στα σύνορα. Στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ασύλου ορισμένες έννοια, έννοιες όπως η έννοια της ασφαλούς ε, τρίτης χώρας δημιουργεί προβλήματα. Η εφαρμογή λοιπόν μιας ε, συμφωνίας επανεισδοχής μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα όταν το πρόσωπο πρόσφυγας δεν είχε πρόσβαση σε δίκαιη διαδικασία ασύλου στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια, μιλάμε για ανθρώπου, οι οποίοι φτάνουν στα σύνορα, δεν του δίνονται η πληροφόρηση που θα έπρεπε για το πώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα ασύλου και απλώ απελάβνονται με εφαρμογή τη συμφωνία επανεισδοχή. κάτι που έχουμε διαπιστώσει σε διάφορε περιπτώσει ε, πρόσφατα σε σημεία ε, των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναφέρω την Λευκορωσία, την, ε, τα σύνορα της Ουγγαρίας αλλά το ακόμα μεγαλύτερο και γνωστό πρόβλημα στη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Πολλοί μιλούν ακόμα και για βίες επαναπροωθήσεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στα... Συζητούνται συμφωνίες επανεισδοχής με την Ουκρανία, με τη Σερβία ή με τη Λευκορωσία και την Τουρκία. Η Ουγγρική Επιτροπή του Ελσίνκη αναφέρει ότι πολύ συχνά πρόσφυγες επαναπροωθούνταν από την Ουγγαρία χωρίς να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, παρόλο που η αστυνομία συστηματικά λέει ότι όλες οι επαναπροωθήσεις έγιναν σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με τις διαδικασίες, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων οι οποίοι ε, απελάθηκαν χωρίς να εξεταστεί ε, καθόλου η κατάστασή τους ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργεί η ε, επιταχυμένη διαδικασία ε, εξέτασης ετοιμάλων ασύλου. Αυτές οι διαδικασίες μπορεί να είναι πολύ μικρής χρονικής διάρκειας και τέτοιου είδους διαδικασίες ε, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται στις συμφωνίε επανεισδοχή με το Μαυροβούνιο, με τη Σερβία, με τη Ρωσία, με την Τουρκία. Το πρόβλημα με αυτές τις επιτυχημένε διαδικασίες είναι ότι αν τελικά ο πρόσφυγα απελαθεί μέσα σε λίγε ημέρε, δεν θα έχει τη δυνατότητα ούτε να ασκήσει έφεση, ούτε να, να, να ασκήσει τα οικονομικά του δικαιώματα, ούτε να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο, ούτε να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία. Με άλλα λόγια, είναι αδύνατη ε, η ε, προσβολή της ε, απόφασης απέλασης. Υπάρχει επίση το ζήτημα της ε, ε, επανεισδοχή και τη επαναπρόθεση ατόμων ε, υπηκών τρίτων χωρών. που συνδέεται και με το πρόβλημα που ήδη σας ανέφερα με την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας. Τι είναι ασφαλής τρίτη χώρα? Μια χώρα η οποία θεωρεί το κράτος μέλος ότι μπορεί να προσφέρει προστασία στον πρόσφυγα και δεν θα ε, κινδυνεύσει εκεί η ζωή του. Έτσι λοιπόν το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διαθέτει το δικαίωμα να επαναπροωθήσει προς μια ασφαλή τρίτη χώρα έναν πρόσφυγα. Η Σερβία για παράδειγμα θεωρείται ασφαλής τρίτης χώρας, τρίτη χώρα, αλλά πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, αποδεικνύουν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί στη Σερβία υπάρχουν πολλά εμπόδια στη διαδικασία ασύλου, το ποσοστό αναγνώρισης είναι σχεδόν μηδενικό, και δεν υπάρχει και καμία δυνατότητα ε, ε, ε άσκησης έφεσης. Τελικά λοιπόν αυτή η έννοια της ασφαλούς τρίτη χώρας υπονομεύει το δικαίωμα του ασύλου. Η εξελόγηση οποιοδήποτε αιτήματο ασύλου θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Θα πρέπει να, να ε, γίνεται αναφορά στις στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε υπόθεση, κάθε προσώπου που ζητάει άσυλο. Και αυτό ακόμα και αν προβλέπεται στον νόμο, στην πράξη δεν ισχύει. Υπάρχει επίση ο κίνδυνο τη αλυσιδωτή επαναπροώθηση, τη απέλαση ενό ατόμου από τη μία χώρα στην άλλη, όπου τελικά καταλήγει σε μία χώρα στην οποία κινδυνεύει η ζωή του και η ελευθερία του. Υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις που έχουν τεκμηριωθεί και δυσμενείς επιπτώσεις ε, μπορεί να είναι τραγικές. Ε, μιλάμε για ανθρώπους που κρατούνται αμέσως μετά την επανεισδοχή τους. Ε, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ουκρανία, για παράδειγμα, μπορεί να βρεθούν στην ίδια φυλακή, με ενήλικες. Όπως είπα, σε πολλές από αυτές τις χώρες προς τις οποίες επαναπροωθούνται άτομα δεν υπάρχουν σωστές ή ούτε καν ε, το απαιτούμενο σύστημα. Η Ουκρανία είναι ε, μια χώρα που δεν διαθέτει ε, αποτελεσματικό σύστημα παροχής ασύλου. Η είπατε του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε μια πρόσφατη της έκθεση τον Ιούλιο καλεί τις χώρες να μην, τις κράτη να μην ε, επαναπροωθούν άτομα προς την Ουκρανία εφαρμόζοντας την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας στο πλαίσιο μιας ε, συμφωνίας, μιας διαδικασίας που έγινε με την Τουρκία, ε, συνήφθη συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία σε μια εποχή που δεν διέθετε αποτελεσματικό σύστημα ασύλου και μάλιστα εφήρμοζε την τακτική, την πολιτική της του γεωγραφικού περιορισμού, δηλαδή περιόριζε τον αριθμό των αιτήσεων ασύλου ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Υπάρχει ένα νέο νομικό πλαίσιο για, την, ε, για το άσυλο στην Τουρκία, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί και ακόμα και όταν ε, υιοθετηθεί θα πρέπει να αξιολογηθεί πρώτα. Η απέλαση, απέλαση λοιπόν προς χώρες ε, transit μπορεί να οδηγήσει στην απέλαση προς την χώρα προέλευσης και τελικά ένα τέτοιο σε μια τέτοια περίπτωση τον άσυλο δεν έχει πρόσβαση. Ένα παράδειγμα θα ήταν η περίπτωση απέλαση ενός προσώπου προς την Ουκρανία που μετά θα απελαθεί προς τη Ρωσία. Από Θα πρέπει λοιπόν τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είναι το πρωταρχικός ε, το πρωταρχικό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζει ένα κράτος μέλος εάν θα συνάψει ε, συμφωνία πανεσδοχής με μια χώρα. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις που τεκμηριώνουν αυτές τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά αυτά είναι μόνο τα περιστατικά που γνωρίζουμε. Είναι πολύ πιθανό ότι τα πραγματικά είναι ακόμα περισσότερα γιατί δεν υπάρχει επαρκής παρακολούθηση, το θέμα ήδη αναφέρθηκε, το θέμα της εποπτείας, δεν θα επανέλθω, αλλά ε, το έκρε καλή και ζητά την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας. Ευελπιστούμε ότι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα έχει την απαιτούμενη διαφάνεια και θα υπάρχει και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για να εξασφαλίσει αυτή τη διαφάνεια. Και ήθε αυτό το πρόγραμμα να μην παραμείνει μόνο ε, ένα πιλωτικό πρόγραμμα περιορισμένης διάρκειας, αλλά να συνεχίσει και μετά. Συμπερασματικά λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις αναφορές για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι αναφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά τη διαπραγμάτευση και κατά την επαναδιαπραγμάτευση ε, συμφωνιών επανεισδοχής. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε μια έκθεση με συμπεράσματα για τις συμφωνίες επανεισδοχής, αλλά δυστυχώς αυτά τα συμπεράσματα δεν υλοποιήθηκαν, δεν υπήρξε συνέχεια που θα έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι σημαντικό το στοιχείο της διαφάνειας, να ξέρουμε τελικά τι γίνεται με αυτές τις συστάσεις. Γιατί όπως σας είπα, οι συνέπειες ε, για κάποιον που απελάβνεται ε, μπορεί να είναι τραγικές και κανείς δεν θα πρέπει ποτέ να απελάβνεται προς μια χώρα στην οποία μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του, η η ελευθερία του, η αξιοπρέπεια του. Και είναι, πιστεύω, και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις τους και να φροντίζει για την αποτελεσματική εποπτεία. Ευχαριστώ. Εμεί σας ευχαριστούμε. Τώρα θα γίνει ο πρώτος γύρος ανταλλαγής απόψεων. Has meeting. Από ό,τι μου λένε δεν ήρθε ο εκπρόσωπος της EEAS, αλλά ήρθε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση HOME. Ναι, αν μου δίνετε το λόγο. Λέγομαι Νίλ Κόλμαν και είμαι πράγματι εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Home που ασχολείται με την επιτήρηση της εφαρμογής των συμφωνιών επανεισδοχής. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν βέβαια είναι πάντοτε πρόθυμες, θα ήταν πρόθυμες να σας κάνουν κοντζάν παρουσίαση σήμερα αν το είχατε ζητήσει γιατί από την προηγούμενη συζήτηση του θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις συμφωνίες επανεισδοχής με το Πακιστάν είχε προταθεί κάτι τέτοιο. Θα κάνω και σήμερα ό,τι μπορώ να σας δώσω μερικές ιδέες. Εμείς παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τις πιθανές επιπτώσεις της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επανεισδοχές και αυτό το βλέπετε σε αρκετή λεπτομέρεια στην αξιολόγηση του 2011 που είχε κάνει η Κομισιόν. Δήλωση μάλλον, όπου ανέφερε και πολλές σοβαρές συστάσεις. Το νομικό πλαίσιο των επανεισδοχών και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σαφές. Πρέπει να τονίσουμε ότι τέτοιες συμφωνίες δεν σημαίνουν ότι τα συμβαλόμενα μέρη μπορούν να μη σεβαστούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Αντίθετα, κάθε φορά επαναλαμβάνεται η υποχρέωση αυτή. Υποχρεώσεις όπως εκείνες που απορρέουν από τη συνθήκη της Γενέβης ή την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων. Τέτοιες συμφωνίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν επί οποιοδήποτε κινδυνεύει να απελαθεί ή να του παραβιαστούν άλλα ανθρώπινα δικαιώματά του γιατί εφαρμόζεται ό,τι έχει απολύτως προβλεφθεί ως εγγύηση για τους ανθρώπους αυτούς. Η Κομισιόν βεβαίως αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ νομικού πλαισίου από τη μία και πρακτικής εφαρμογής από την άλλη και γι' αυτό στην αξιολόγηση του 2011 που ανέφερα και προηγουμένως κάναμε ορισμένες συστάσεις για την εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων. Μερικά από αυτά τα συνοδευτικά ή παράπλευρα μέτρα θα τα δείτε στις τελευταίες συμφωνίες επανεισδοχών που διαπραγματευθήκαμε και πρόσφατα η Επιτροπή ΕΛΕΦ, ΛΥΜΠΕ δηλαδή, ε, συζήτησε την σχετική συμφωνία με την Αρμενία που θα, θα ψηφιστεί στις 9 Οκτωβρίου. Είναι η πρώτη τέτοια συμφωνία, θα το δείτε, που έχει νέες ρήτρε ε, και εγγυήσεις. Ένα πρόσθετο άρθρο δηλαδή για το σεβασμό των συμβαλωμένων μερών ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδίως της χώρας που δέχεται τον επανεισδεχόμενο και επίσης για πρώτη φορά υπάρχει κάτι καινούριο, δηλαδή η δυνατότητα να παγώσει η συμφωνία αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Εκτός αυτού η Κομισιόν επιτηρεί, παρακολουθεί το μελλοντικό της πρόγραμμα εφαρμογής τέτοιων επανεισδοχών στην Ουκρανία και το Πακιστάν. Πειραματικά θα το παρακολουθούμε τρία χρόνια γιατί θέλουμε να είναι όλα πολύ διαφανή. Με συνεργασία και της υπάτης αρμοστίας του ΟΗΕ και μήκη όμικρον. Για να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει πρακτικά. Αυτό βέβαια προστίθεται στην αξιολόγηση και επιοπτία που ήδη γίνεται κανονικά και με τις προηγούμενες συμφωνίες επανεισδοχής. Τέλος, για την επανεισδοχή πολιτών τρίτων χωρών, δηλαδή ούτε της μίας ούτε της άλλης συμβαλόμενης χώρας τέτοιου είδου επανεισδοχέ μα ανησυχούσαν ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα επί πολύ καιρό και θα έπρεπε να σημειώσουμε ότι συνήθω τέτοια ρήτρα χρησιμοποιείται πάρα πολύ σπάνια. Στα εξωτερικά σύνορα με την επιταχυμένη διαδικασία μπορεί να υπάρξει η περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας που να, επαν, που να τύχει επανεισδοχής, αλλά επειδή είναι σπάνιο δεν το έχουμε ακόμα εξετάσει, μπορεί να χρειάζονται και εδώ βελτιώσεις και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν στο μέλλον. Χρειάζεται να γνωρίζουμε τα πράγματα πληρέστερα, γενικότερα για τις επανεισδοχές, αλλά ιδίως για πολίτες τρίτων χωρών. Περισσότερα και ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα θα μας βοηθούσαν πολύ για να γίνονται συζητήσεις σαν τη σημερινή. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Η συμπρόδο. Λοχμίλτερ θα έχει τον τελικό λόγο για να κάνει τα συμπεράσματά της στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε ε, εμπειρογνώμονες. Εγώ λυπάμαι που δεν είναι κανείς εδώ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης γιατί τους είχαμε ζητήσει να είναι εδώ και θα είχε, όπως είπε και ο κύριος Κασαρίνο, προστιθέμενη αξία το να εστιάσει η ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της προσπαθία της και σε αυτόν τον τομέα. Θα σας θέσω ορισμένα ερωτήματα τώρα. Ελπίζω ότι είναι εύστοχα τα ερωτήματα αυτά. Είπατε ότι υπάρχει μια κοινή επιτροπή επανεισδοχής η οποία ασχολείται με τα τεχνικά θέματα. Και τώρα <clears throat> άκουσα και από όλους τους ομιλητές ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει πιο ανεξάρτητη παρακολούθηση αυτών των θεμάτων. Κατά την άποψή σα λοιπόν πώ θα έπρεπε να γίνει αυτή η παρακολούθηση στην Κοινή Επιτροπή επανεισδοχή, Θεωρείτε ότι λειτουργεί αυτό ήδη ή χρειάζεται περισσότερη παροχή ανεξαρτήτων εκθέσεων. Δεν θέλω τώρα να <clears throat> είμαι προκατηλημένη. Αλλά από το παρελθόν έχουμε διδαχθεί ότι μόνο όταν υπάρχει σαφή τεκμηρίωση από ανεξάρτητες μήκη ο για το τι έγινε με τα άτομα τα οποία ε, ήταν αντικείμενα επανειστοχής. Μόνο τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιδράσει στα θέματα αυτά. Υπάρχει μια περίπτωση που εμπλέκει την Ιταλία στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όταν απεστάλησαν κάποια άτομα στην Λιβύη του Καντάφη, ήταν θύματα βασαναστηρίων και μόνο με τη βοήθεια των ΜΚΟ υπήρξε η δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο του Στρασβού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η λήψη μιας απόφασης υπέρ τους. Ξέρουμε ότι τώρα υπάρχουν και κάποια συνοδευτικά στοιχεία διασφάλισης <clears throat> για να κάνουμε πιο πρακτικό το νομικό πλαίσιο. Θα ήταν χρήσιμο όμως από τη δική σας πλευρά να μας πείτε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την παρακολούθηση για τις υποθέσεις αυτές είπατε μετά ότι η Σερβία δεν είναι ασφαλής χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την κατάσταση στη Σερβία και να στείλουμε ίσως και μια αντιπροσωπεία και να εξετάσουμε το θέμα αυτό πιο προσεκτικά. Οι διαδικασίες ασύλου ή το δίκαιο ασύλου στη Σερβία είπατε ότι το κριτήριο τα κριτήρια για την ε, επαρισδοχή θα πρέπει να μπορούν να τύχουν μιας προσφυγής. Όχι, όχι, λέει, πρέπει να ενημερωθούν, λέει ο κύριος Κασαρίν. Τώρα πια πρέπει να κάνουμε μια επανεξέταση. Εντάξει, ωραία. Για την κυρία Σιράμα, για την εποπτεία. Μιλήσατε για τα πιλωτικά προγράμματα που σχεδιάστε να υλοποιήσετε. Έχετε ήδη υφιστάμενες <clears throat> περιπτώσεις όπου προσέφυγαν οι ενδιαφερόμενοι στα δικαστήρια γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν απέσταλσαν στην χώρα προέλευσής τους ή σε μια τρίτη χώρα. Ίσως να μαζέψουμε τα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Και στο Ίκρε θέλετε να έχετε πιο ισχυρές διασφαλίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπα ότι πρέπει να υπάρχει καλή νομοθεσία στις αρμόδιες χώρες και αναφερθήκατε επίσης και στους μηχανισμούς παρακολούθησης και εποπτείας. Έχετε περαιτέρω κριτήρια. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αναστέλλεται η εφαρμογή των συμφωνιών επανιστοχής, mm. κατά την άποψή σας. Σε τι χώρες λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσετε αυτή η αναστολή των συμφωνιών επανεισδοχής. Αυτά από μένα. Για να ταξινομήσουμε και να τακτοποιήσουμε τον γύρο των απαντήσεων στα σχόλια, τις απόψεις, τις συστάσεις των λεγόμενων της Προέδρου πρότεινε να το δώσουμε λόγο της κυρία <clears throat> Ρομέρο Λόπεθ, η οποία θέλει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις και αν υπάρχει κάποιο άλλο μέλος το οποίο θέλει να λάβει το λόγο, παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε τις ερωτήσεις και να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας για την ευκαιρία να που είχαμε να πληροφορηθούμε από αυτούς για τις συμφωνίες αυτές επανεισδοχής και επίσης επειδή είναι παρούσα και η Κομισιόν <clears throat> θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε περισσότερο λεπτομεριακά για τις περιπτώσεις όπου τίθεται σε εφαρμογή η οδηγία περί επιστροφής γιατί αυτή η οδηγία μπορεί να έχει μεταγραφεί σε διάφορες χώρες με διαφορετικό τρόπο. Ο χρόνος κράτησης, οι συνθήκες κράτησης και όλα αυτά ποικίλουν από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα της Κομισιόν το 2011 σε σχέση με τα θέματα αυτά ανέφερε ότι πρέπει ορισμένε πτυχές των συμφωνιών επανεισδοχής να επαναξεταστούν και ορισμένα στοιχεία αυτή τη οδηγία για την ε, ε, επανα, επαναφορά των ε, μεταναστών δεν μας φαίνονται απόλυτα σύμμορφες με, την, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Κομισιόν θα έπρεπε να μας εξηγήσει γιατί μπορούν να υπάρχουν τόσο διαφορετικά διαστήματα κράτησης για αυτούς οι οποίοι είναι αιτούντες άσυλο και για τους παράνομους μετανάστες επίσης και γιατί <clears throat> δεν υπάρχουν ε, παρεμβάσεις για να καταγγελθούν αυτές οι κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων σε πολλές χώρες. Θα ήταν χρήσιμο εμείς λοιπόν ως κοινοβουλευτικοί να έχουμε πληροφόρηση για τα θέματα αυτά για να μπορέσουμε να καταγγείλουμε αυτή την κατάσταση και να εξασφαλίσουμε μια πιο ανθρώπινη μεταχείριση ατόμων που δεν έχουν διαπράξει κανένα δίκημα, απλώς είναι κρατούμενοι λόγω διοικητικών ε, ελλείψεων και παράνομης εισόδου. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας κάνω μία πλοϊκή ίσως ερώτηση, κυρία Πρόεδρος. Ε, το έθεσε λογικά, αλλά παρόλα αυτά. Με παραξένεψε οι δηλώσει δύο εμπειρογνωμόνων που είπαν ότι η Σεριβία δεν είναι λέει ασφαλής χώρα. Ω Θεέ μου, μα πώς μπορεί, θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε ρεαλιστικά όμως. Πριν από δύο χώρες, ο, χρόνια χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έτυχαν απελευθέρωσης των θεωρήσεων για να επισκέπτονται το χώρο του Σένιγκεν. Άμα δεν είναι ασφαλής χώρα, πώς μπορούν οι Σέρβοι να κυκλοφορούν χωρίς βίζα. Ζητάνε πολιτικό άσυλο πολλοί Σέρβοι. Για πέστε μου. Αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τέθηκε ένα ερώτημα στην Κομισιόν και μετά οι εμπειρογνώμονες. Μήπως ο κύριος Κόλμαν θέλει να απαντήσει σε αυτά που σας είπε ο κύριος Ρωμέρο Λόπεθ. Κυρία. Η κυρία, η κυρία, κυρία. Όχι, αλλά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου εδώ εξ αριστερών. Καλησπέρα σας. Από το ερώτημά σας κατάλαβα ότι αναρωτιέστε γιατί οι κανόνες που ισχύουν για τις επανεισδοχές δεν γίνουν, έχουν τύχει πλήρους εναρμόνισης, δεν είναι οι ίδιοι σε όλες τις χώρες. Μα αυτό είναι ακριβώς το πνεύμα των επανεισδοχών να υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας. Τώρα για τις κρατήσεις υπάρχουν πολύ σαφείς όροι και κανόνες και οι σχετικές διαπραγματεύσεις υπήρξαν πολύ δύσκολες για να υπάρξει σεβασμός των δικαιωμάτων. Τα κράτη-μέλη χρειάστηκε να δεχτούν ότι η κράτηση παραδείγματο χάρη είναι τελευταίο μέτρο. Και βέβαια δεν έχουμε ακόμη πλήρως εναρμονισμένα συστήματα και τις ίδιες περιόδους κράτησης. Μπορεί αυτό να μην τις ικανοποιεί όλους, αλλά αυτά που πετύχαμε με την οδηγία είναι ήδη ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ιδέα αξιολόγηση για τη μεταφορά της οδηγίας στις χώρες μέλη ακόμη συνεχίζεται και ως θεματοφύλακ των συνθήκων εμείς, ε, η Κομισιόν δηλαδή, εξετάζει όλες τις λεπτομέρειες. Αν υπάρχουν δεδικαιολογημένες περιπτώσεις για εξαιρέσεις θα τις δεχτούμε. Ωραία. Τώρα οι ομιλητέ. Η κυρία Λοχμπίλερ νομίζω έθεσε μερικά ερωτήματα. Είπα έχουμε χρόνο και για δεύτερο γύρο και μετά θα λήξουμε. Λοιπόν. Ποιος θα μιλήσει πρώτος, μήπως η κυρία Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις που θέσατε κύριε Λόχπιλε. Η πρώτη είναι γιατί αυτή η εποπτεία είναι πιο τεχνική και όχι περισσότερο εστιασμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι κοινέ επιτροπές ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, χωρών με τις οποίες υπάρχουν ε, συμφωνίες επανεισδοχής είναι απλώς πολυμερείς επιτροπές, επιτροπές στις οποίες γίνεται συζήτηση μεταξύ των μερών που έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία επανεισδοχής. Επομένως τελικά πώς θα μπορούσαν να είναι ουδέτερες και ανεξάρτητες. Γίνεται μια τεχνική συνεννόηση, πόσο γρήγορα πρέπει να ε, υπάρξει απάντηση κάθε φορά που υπάρχει αίτημα επανεισδοχής, τέτοιου είδους συζήτηση. Ή επίσης πώς θα φροντίσει η χώρα προς την οποία γίνεται η επανεισδοχή για τα ε, άμεσες ανάγκες ε, του αναπροεθούμενου. Και για να έρθει και στο δεύτερο ερώτημά σας για την εποπτεία, όταν εντοπίστηκαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσωπικά έχω ασχοληθεί με το ζήτημα της Ουκρανίας και μαζί με την υπατερμοστία και το ΕΚΡΕ δημιουργήσαμε ένα εργαλείο. Ονομάζεται το, το ο μηχανισμός παρατή, ε, εποπτείας ε, πριν λίγα χρόνια και προσπαθεί να εξετάζει το κατά πόσον οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες ε, και στα δικαιώματά τους. Και ανάμεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που απεστάλησαν από χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με συμφωνία πανεσδοχής. Και αυτό που διαπιστώσαμε με αυτό το παρατηρητήριο είναι ότι πρόσφυγε οι οποίοι υπέβαλαν έτοιμη ασύλου σε χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εστάλησαν στην Ουκρανία. Η Ουκρανία θεώρησε ότι αυτό αρκεί, δεν, αυτή τη στιγμή εξετάστηκε το αίτημά του και απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται η Ουκρανία να το εξετάσει. το δικαίωμα ε, να έχει κανείς πρόσβαση σε δικηγόρο, σε διερμηνέα, να αντιληφθεί την ε, διαδικασία που γίνεται στο Ουκρανικά, να έχει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Δεν γίνεται σεβαστό, αλλά νομίζω ότι με το διάλογο και με τη συνεργασία με τις Ουκρανικές αρχές καταφέραμε πολλά. Αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα και η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Κύριο Κασαρίνο, θα προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω στις ε, ερωτήσει που μου απευθύνατε. Τώρα για την Κοινή Επιτροπή Επανεισδοχών, για κάθε συμφωνία επανεισδοχή δημιουργείται μια τέτοια επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς από τις δύο χώρες που έχουν συνάψει, ε, μάλλον από τη χώρα που, έχουν, που έχει συνάψει την Συμφωνία Επανεισδοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσώπους του κράτους μέλους. Αλλά δεν συνεργάζονται όλα τα κράτη-μέλη διμερώς με μια τρίτη χώρα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας επανεισδοχής επί τη βάση ενός εφαρμοστικού πρωτοκόλου. Θα έλεγα ότι δεν είναι συνεκουανόν. Αυτό δεν είναι προαπαιτούμενο. Από τις Κάποια από τα κράτη-μέλη δεν έχουν συνάψει τέτοιο εφαρμοστικό πρωτοκόλλο και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί από τη στιγμή που υπάρξει αυτή η ρήτα, υπάρχει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, τα πράγματα διασαφηνίζονται. Mm. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Αλλά δυστυχώς όπως σας είπα, δεν συμβαίνει πάντα με όλες τις συμφωνίε επανεισδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνα το πλαίσιο είναι διαφορετικό. Τώρα πια έχει ενισχυθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της συνήθω νομοθετική διαδικασία. Κατά την άποψή μου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ακόμα και την παρακολούθηση του πώς εφαρμόζονται αυτές οι συμφωνίες επανεσδοχής. Ε, ελπίζω μια μέρα να το δούμε και στην πράξη όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να, να, να αναλάβει τις ευθύνες του το Κοινοβούλιο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης είναι το, το ζήτημα πώς θα επιλεγούν οι τρίτες χώρες με τις οποίες θα συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνία Πανεσδοχή. Και σε αυτό έχει τη δυνατότητα να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να γίνονται αυτές οι επιλογές με σαφή κριτήρια. Ελπίζω να απάντησα. Σερβία. Όχι, η Σερβία δεν είναι ασφαλή τρίτη χώρα. Θα αναφερθώ στην έκθεση που δημοσιοποίησε πέρσι, το 2012, η τη Αρμοστέα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Πιστεύω ότι αν μη τι άλλο οι εκθέσεις της ΥΠΑ ΕΕ της είναι σοβαρές. Έχουν γίνει μετά από σοβαρή αξιολόγηση και μπορούν να διαφωτίσουν εκείνους που χαράζουν πολιτικές. σε μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της, του 2005 για τη διαδικασία ε, για, για το άσυλο. Στο άρθρο 27 ορίζεται επακριβώς η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας. Μπορώ να σας το στείλω αυτό το έγγραφο για να δείτε ποια είναι τα κριτήρια, εκεί καταγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια. Ευχαριστούμε. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Το πρώτο ερώτημα είναι για τη ρήτρα αναστολής. Είναι σημαντικό αυτό και υπήρχαν και κάποιες ε, συστάσεις σχετικά με την Κομισιόν. Αν έχετε ήδη μια διασφάλιση σε μια συμφωνία που λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η και τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχετε μία μνήα όλων των συμβάσεων και των συμφωνιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει. Μας βοηθάει αυτό για τη χώρα που υπάρχει η επενδοχή. Μας λένε τώρα ότι η Σερβία ή το Πακιστάν ή η Σερβία ή η σερβια η η τουρκια δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. αν υπάρχει μια οποιαδήποτε παράνομη κράτηση ή παραβίαση δικαιωμάτων, αν τα άτομα κρατούνται συστηματικά όταν γυρίζουν και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα δικαστικής προσβολής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό είναι μια παραβίαση των δικαιωμάτων τους, είναι παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν τους κακομεταχειρίζονται αν η κατάσταση στη χώρα αυτή είναι τόσο δύσκολη και τόσο άσχημη ώστε υπάρχει κακομεταχείριση. Μπορείτε να σκεφτείτε την υπόθεση του Βελγίου με την Ελλάδα που είπε το δικαστήριο ότι θα θεωρηθεί το κακομεταχείριση αν τους στέλνανε πίσω αυτούς τους ανθρώπους στην Ελλάδα και εδώ μιλάμε για την Ευρώπη. Επρόκειτο λοιπόν για ήδη μεταχείριση που ισοδυναμούσε με κακομεταχείριση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν <clears throat> καταγράφονται αυτά τα θέματα. Θα πρέπει τότε να ανασταλεί η Συμφωνία Επανεισδοχής και αν μας λένε οι εκθέσεις ότι η Ουκρανία δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η Συμφωνία Επανεισδοχής για χώρες όπως η Ουκρανία. Και για να επαλέθω ότι είναι μια ασφαλής χώρα. Μιλάμε τώρα σε επίπεδο νομικό. Όχι, η Σερβία δεν είναι ασφαλής χώρα. Για τους ετούμενους ασύλου μπορεί για ένα Σέρβο τον ίδιο να μην είναι ασφαλής η χώρα. Χρειάζονται πολλές φορές άτομα τα οποία Υπάρχουν άτομα τα οποία πολλές φορές διώκονται στο ίδιο του το κράτος και μπορούν να ζητήσουν άσυλο σε άλλες χώρες. Την πρώτη οδηγία για άσυλο περιλαμβανόταν και η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει ένα κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να γίνει γιατί δεν συμφώνησαν ποτέ για αυτό τον κατάλογο. Τι είναι ασφαλής μια χώρα είναι κάτι που δεν ξέρει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη. Η Σερβία και άλλες χώρες δεν είναι μέσα στον κατάλογο των ε, ασφαλών χωρών. Το αν είναι ασφαλής ή όχι μια χώρα εξαρτάται από το συγκεκριμένο άτομο. Και δημοσιεύσαμε μια έκθεση με τις πληροφορίες που έχουμε και έχουμε ε, μαρτυρίες ετούντων ε, ασύλου και μεταναστών. Μια γυναίκα από, την, ε, από το Αφγανιστάν η οποία τώρα βρίσκεται στην, Ουγγαρία και της δόθηκε προστασία. Ε, πίσω στο σύνορο της Σερβίας στη μέση του χειμώνα, την αφήσαν στην άλλη άκρη σύνορων στο χιόνι κατάφερε να γυρίσει στην Ουγγαρία επειδή ήταν νέα και ανθεκτική και κατάφερε να πάρει το καθεστώς του ετούντος ασύλου στην Ουγγαρία. Λοιπόν, στην Σερβία δεν είχε καμία δυνατότητα αποστασίας και πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Ευχαριστώ, δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει να λάβει το λόγο. Δεν βλέπω κάποιον ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο, κάποιο εκπρόσωπο οργανισμού, Εάν είναι έτσι τα πράγματα λοιπόν, νομίζω ότι φτάνουμε στα συμπεράσματα αυτής της ε, συνεδρίας και ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάλει. Και τώρα, κυρία Συμπρόεδρε, κυρία Λόχιλα, θέλετε να λάβετε το λόγο. Ναι, και εγώ μπορώ να κλείσω με μια ωραία παράθεση. Mm. Ε. Και καλό που κάναμε μαζί αυτή την ακρόαση. καταγράφω από την πλευρά της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα λεχθέντα και θα ήθελα να ακούσω και στο μέλλον από, την, από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ποια είναι τα πορίσματα της, ε, των πιλωτικών προγραμμάτων. Όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στην έκθεση στην ενδιάμεση για το πρόγραμμα ε, της Στοκχόλμης και έχω αυτό το οποίο σας λέει ένας συνάδελφος για αυτή την Επιτροπή τη Μικτή Επιτροπή Επανεισδοχής, λέει ζητούμε από την Επιτροπή να επιτρέψει όχι μόνο το Κοινοβούλιο, αλλά και ο να συμμετέχουν στην ε, Κοινή Επιτροπή Επανεισδοχής και να παροτρύνουμε την Κομισιόν να δώσει το Κοινοβούλιο πρόσβαση στα έγγραφα που προετοιμάζει αυτή η Επιτροπή. Είναι η ελπίδα μας λοιπόν ότι η Επιτροπή Λίμπε και η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν σε αυτή τη σύσταση γιατί αυτό θα βοηθήσει να βελτιωθεί το έργο αυτής της κοινή Επιτροπής Επανεισδοχής γιατί μετά από αυτά που λέμε με την περίπτωση που αναφέρατε στο τέλος νομίζω ότι είναι πολύ συχνό αυτές οι πολιτικές αντιμετώπισης των προσφύγων και ατόμων που επαναπροωθούνται <clears throat> είναι σκανδαλώδης κατάσταση και μόνο με ένα τέτοιο σκανδαλώδης γεγονός μπορεί να πιστούν η πλειοψηφία των βουλευτών να αλλάξουν τις πολιτικές. Αν δεν υπάρχει λοιπόν καμία βοήθεια προς τα άτομα αυτά, θα πρέπει να επαναξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Δυστυχώς δεν έχουμε μια πολιτική για τους πρόσφυγες που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και σας ευχαριστώ που ήρθατε και συμπροεδεύσατε μαζί μου. Πολύ το χάρηκα και εγώ λέει ο κύριος Λόπες Αγγιλά. Σας ευχαριστώ όλους. So those colleagues for, um, from I have to remind you that tomorrow we meet in a different room. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα συναντηθούμε σε άλλη αίθουσα. ASP 3G3. Ευχαριστώ.